Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω τι κάνουμε τόση ώρα, κύριε Πρόεδρε. Το, δικό μου το ρολόι δείχνει 10 και 10. Η ώρα περνάει. Ε, με ενημέρωσαν πως κάποιοι συνάδελφοι ακόμη προσπαθούν να έρθουν. Α, εντάξει, θα να μην περιμένουμε άλλο. Άρχεται η συνεδρίαση, σας καλωσορίζω όλους. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή, κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν θα, πληρώσουμε, ε, ψηφίσουμε την έκθεση Βλάσακ, απλά θα έχουμε μια ενημέρωση. Ε, Βεβαίω μεταδίδεται και στο διαδίκτυο η συνεδρίαση. Όπως ξέρετε, περνάμε στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης, έγκριση των πρακτικών της 24ης 24 ε, Νοεμβρίου τα οποία τα έχετε και αν μέχρι το τέλος συνεδρίασης δεν υπάρχει αντίρρηση, θεωρείτε ότι εγκρίνονται. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε, περνάμε στην ψηφοφορία. Ναι, κύριε Πίπερ. Μετά κυρία Σρέντερ. Ο Μάρκος Πίπερ. Παρακαλώ. Περιμένετε λίγο να βάλω τα ακουστικά μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω πει επανειλημμένος πως δεν συμφωνώ με την καθυστέρηση στο θέμα της μακροοικονομικής αρεσιμότητας και θα πρέπει φοβάμαι να απόσχομαι από την ψηφοφορία γιατί από ό,τι φαίνεται θα περάσει να συμφωνήσουμε σήμερα σε κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί 100% το Συμβούλιο. Πρόκειται για τη λέξη persistent, δηλαδή για μια διαρκή και μόνιμη ε, ε, αναβολή ε, της ε, ε, κατάστασης και θα πρέπει να περάσουμε 5, 6, 7 εμπόδια για να υπάρξει μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Δηλαδή δεν θα έρθει ποτέ. Πολύ απλά. Οπότε σας παρακαλώ να προσέξετε πάρα πολύ εδώ πέρα με τη σημερινή ψηφοφορία ρισκάρουμε δεύτερη ανάγνωση κυρία Πρόεδρε αν προστίθενται λέξεις που δεν τις έχουμε διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο. Είτε λοιπόν η λεξούλα αυτή persistent, μόνιμη, φεύγει, αλλιώς εγώ δεν μπορώ να συμμετάσχω στην ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, αυτό δεν ε, έχει σχέση με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Εάν έχετε κάτι να πείτε για την έκθεση ε, ε, Εκεί πέρα βρισκόμαστε. Αν όχι, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο στο οποίο αναφέρεστε. Λοιπόν, να ξεκινήσει η ψηφοφορία για την έκθεση Γιάνν Όλμπριχτ ε, για την ε, επί της διαδικασίας. Μα ήταν μια παρατήρηση επί της αρχής, λέει ο κύριος Πίπερ. Είχα την αίσθηση πως θα ε, ξεκινήσετε και δεν θα επιτραπούν άλλες δηλώσεις. θα ξεκινήσετε την ψηφοφορία, γι' αυτό έκανα τώρα την δήλωση αυτή. αυτό και θα ήθελα απλά να αναφερθεί, να σημειωθεί πως αναφερόμουν στον γενικό, στη γενικότερη κατάσταση. Πρόεδρος. Καλά, καλά, δεν ξέρω τι θέλετε εσείς, εγώ ξέρω, ξέρω πάντως ότι θέλω να τα βρούμε και να τα συζητήσουμε. Μάρκος, ε, θετικά βλέπω τα πράγματα, οπότε για να ξεκινήσουμε τώρα με την ε, ψηφοφορία επί της έκθεσης Όλμπρεχτ. Ελισάβετ, εάν δεν είναι για την έκθεση Άλμπριτ, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την ε, ψηφοφορία για αυτή την έκθεση. Αν θες κάτι να πεις για μια άλλη έκθεση, ε, για την οποία συζητήσουμε αργότερα, να το κάνουμε αργότερα. Οπότε σε παρακαλώ, ας ε, αρχίσουμε, ας ακολουθήσουμε την μεσία Οπότε αρχίζουμε την ψηφοφορία. Άμε με, με, με αναστάτωσαν αυτά που είπε ο Μάρκος και ξέχασα να βγάλω έξω την ηλεκτρονική κάρτα. Οπότε, για να κάνουμε πρώτα πρώτα μία ε, δοκιμή να δούμε αν δουλεύουν τα μηχανήματα. Ψηφίζουμε. Κάποιος δεν ψήφισε. Αλλά δεν έχει σημασία από ό,τι φαίνεται ολονών τα μηχανήματα δουλεύουν. Και άρα συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Το, η τροπολογία υπάρχει μόνο δύο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε πάμε τώρα στο σύνολο της νομοθετικής πρότασης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε Πέρας. Και έχουμε 35 υπέρ, επομένως εγκρίνεται. Και επίσης τώρα την νομοθετική πρόταση ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται. Και τώρα για τις διοργανικές διαπραγματεύσει. Χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 38-1. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, τώρα πάμε στο επόμενο σημείο που είναι το 6 στη μέση και που αφορά κάποιους ε, κανονισμούς. Οπότε ξεκινώ με ενημέρωση. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κωδικοποιημένου κειμένου το οποίο το έχετε λάβει χθε. Αυτό περιλαμβάνει την έκθεση που ψηφίσαμε στην Επιτροπή τον ε, Ιούλιο φέτος. Επίσης, θα ψήσουμε το τέλεσμα των ε, διοργανικών ε, διαπραγματεύσεων όπως έλαβαν χώρα στη συνέχεια. Οπότε και αυτό είναι το αποτέλεσμα του τριμμένου διαλόγου όπως έγινε στο Στρασβούργο. Και αυτά τα οποία σήμερα θα ψηφίσουμε θα περιλάβουν και τις διατάξεις αυτές στις οποίες αναφέρθηκε ο Μάρκος Πίπερ. Να δώσουμε στον Φανή ε, λόγο που είναι ασυγητής και κατόπιν στην συνεισηγήτρια. Ε, την Κωνσταντς. Ναι, αλλά να να το κάνουμε σύντομα. Γιατί τα έχουν πει τόσες φορές, οπότε απλώς να κάτσουμε να δούμε τα τελευταία αποτελέσματα. Αυτά δηλαδή που αποσπάσαμε. Τόσοι και τόσοι τριμμένες διάλογοι, τόσες διαπραγματεύσεις, άρα εγώ θα ήθελα σήμερα να ψηφίσουμε. Και να μπορέσουμε να απεμπλέξουμε το σύριαλ του MFF του πολιετούς πλαισίου. Όλα βρίσκονται στην έννοια που έχετε λάβει. Για μένα όσο πιο γρήγορα προχωρήσουμε τόσο καλύτερα. Κωνσταντία, πριν λάβεις το λόγο, ε, θέλει ένα διαδικαστικό η Ελισάβετ. Για πέστε μας. Προσπάθησα πολλές φορές ε, εγκαίρως ε, να πω πως έχω κάτι για να μπει στην ημερήσια διάταξη. Αναβλήθηκε Μα όταν έχουμε ένα τέτοιο σημείο, σας παρακαλώ να, να εισακούγεται. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ πέρα, με ποια βάση ψηφίζουμε. Δεν υπάρχει κατάλογος ψηφοφοριών που να έστειλε η γραμματεία. Τίποτα τέτοιο. Δεν είχαμε δυνατότητα να υποβάλουμε τροπολογίες και χωριστές ψηφοφορίες. Αλλά ο κανονισμός μας ε, το επιτρέπει αυτό για ε, ψηφοφορίες στην Επιτροπή. Δηλαδή και χωριστές ψηφοφορίες και τροπολογίες το επιτρέπει. Και έχουμε επανειλημμένως ζητήσει κατάλογο ψηφοφοριών και τη δυνατότητα αυτή μας λέτε πως δεν γίνεται. Κατά την άποψή μου εδώ πέρα παραβιάζεται ο κανονισμός. Θέλω να μάθω λοιπόν με ποιο, ε, πού βασιζόμαστε στον κανονισμό και διεξάγεται ψηφοφορία. Ε, έπρεπε... Σε, σε ποιο άρθρο αναφέρεστε. Ε, έπρεπε να το έχετε πει όταν ζητήσατε το λόγο επί της διαδικασίας. Δεύτερον, ψηφίζουμε σήμερα επί του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχει άρα κατάλογος ψηφοφοριών σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό δεν τον λάβατε. Θα έχετε δυνατότητα να προετοιμάσετε τροπολογίες και χωριστές ψηφοφορίες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για την Ολομέλεια. Αλλά τώρα είμαστε εντός του κανονισμού, τον οποίο έχουμε ελέγξει πολλάκι. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αυτή ήταν η απάντησή μου. Ναι, παρακαλώ. Ε, εγώ βασίζομαι στο άρθρο 70, όπου δεν αποκλείεται η δυνατότητα υποβολής ε, τροπολογιών ε, ούτε στο πλαίσιο της πρώτης ανάγνωσης. Είναι σαφές. Δεν αποκλείεται. Σαφώς. Οπότε έπρεπε να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ή τουλάχιστον εγκαίρος να μας ε, τουλάχιστον να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πως δεν συμφωνούμε με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα υπό τη μορφή που έχει και να ζητήσουμε τροπολογίες και χωριστές ψηφοφορίες. Η νομική γνωμοδότηση είναι διαφορετική. Θα σας παρακαλέσω να δείτε το άρθρο 70 ε, εδάφιο 5, όπου δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Τέλος πάντων, είναι διαφορετική η ερμηνεία του κανονισμού. Θα ήθελα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Άλλα σχόλια επί της διαδικασίας. Εάν όχι... Α, με συγχωρείτε κυρία Ένστ. Επί της διαδικασίας φαντάζομαι. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέει η κυρία Σρέντερ. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω η πτυχή αυτή της ε, μακροοικονομικής αιρεσιμότητας τουλάχιστον να είναι χωριστή ψηφοφορία. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω για όλες τις ε, πολιτικές ομάδες. έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον να ξεκαθαρίσουμε την ε, στάση μας μέσω χωριστής ψηφοφορίας. Δεν ξέρω σε ποιο άρθρο βασίζεστε. Φαντάζομαι. Επί της διαδικασίας μόνο παρακαλώ. Κύριε Σούκες, πείτε μας όμως το άρθρο στο οποίο αναφέρεστε. Μάλιστα, Πρόεδρε. Εγώ επικαλούμε το άρθρο 70, ώστε να ζητήσω να κάνουμε διαφορετική ψηφοφορία. Γιατί εδώ ψηφίζουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην συνεννόηση με, όσον αφορά την διοργανική συμφωνία. Ενώ δεν θα πρέπει να αρνούμεθα ότι στην ουσία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό της ε, Επιτροπής μας για ορισμένους τομείς και ιδιαίτερα για την μακροαιρεσιμότητα. Εγώ, αν ε, ε, ψηφίσουμε, είμαι υποχρεωμένος να καταψηφίσω την διοργανική συμφωνία. Αλλά δεν θέλω να φανώ ότι είμαι κατά του ορισμού κονδυλίων γρήγορα, αλλά με αναγκάζεται να ψηφίσω κατά. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την Επιτροπή μπορούμε να ψηφίσουμε με μία τροπολογία μεμονωμένου βουλευτή, ενώ στην Ολομέλεια πρέπει να βρούμε τουλάχιστον 40 ε, βουλευτές για να υποβάλουμε τροπολογία. Οπότε δεν είναι άσχετο το θέμα. Γι' αυτό ζητώ να προχωρήσουμε μέσω μιας διάκρισης επί της ουσίας πριν να μπορέσουμε να δώσουμε την έγκριση στην διοργανική συμφωνία. Συνάδελφοι, καταλαβαίνω πως ερμηνεύετε διαφορετικά τα πράγματα, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω σαφώς πως αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μία ψηφοφορία. Υπέρ, κατά και αποχή. Την έκθεση την ψηφίσαμε τον Ιούλιο. Σήμερα ψηφίζουμε επί το αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων, όπως αυτό ε, φαίνεται στο ενοποιημένο κείμενο. Ε, Ελίζα Μπεθ, άφησε με να τελειώσω. Δεν σας διέκοψα. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα τον κανονισμό. Αυτό το οποίο μπορούμε να έχουμε σήμερα είναι μία μόνο ψηφοφορία. Α, λοιπόν, έτσι, έτσι έχει η διαδικασία, μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει πως ε, σας εμποδίζει κανείς να κάνετε ό,τι θέλετε και να προτείνετε χωριστή ψηφοφορία ή οτιδήποτε άλλο για την Ολομέλεια. Αλλά στην Επιτροπή την ψηφίσαμε ήδη την έκθεση. Δεν θα την ξαναψηφίσουμε. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Ελίζαμπεθ. Ναι, επί της διαδικασίας πάλι από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Εμείς αναφερόμαστε στο άρθρο 70. Αυτό είναι το σχετικό άρθρο. Είναι σαφές. Και εκεί πέρα δεν αποκλείεται η δυνατότητα χωριστής ψηφοφορίας και τροπολογιών. Δηλαδή επιτρέπεται. Και είναι σαφές πως δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε κάποια στιγμή στο παρελθόν. Είχαμε ψηφίσει και η θέση του Κοινοβουλίου ήταν απόρριψη της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Τώρα μας προσφέρεται εδώ πέρα ένα αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που είναι σαφής έγκριση της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Υπάρχει η δυνατότητα να το ψηφίσουμε χωριστά και ετούμε το άρθρο 21 και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για το άρθρο 21 και το άρθρο 19 να ψηφιστούν ξεχωριστά. Και επίσης ετούμε να διαγραφούν αυτά τα δύο άρθρα της Κομισιόν. Αυτά νομίζω εγώ πρέπει να ψηφίσουμε για να επανέλθουμε στην εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βεβαίως είναι δικαίωμα της ε, Επιτροπής να επανέλθει στο, στην εντολή του Κοινοβουλίου. Δηλαδή να βάλει ένα πλήν να πει όχι στην μακροοικονομική ρεσιμότητα. Γι' αυτό χρειάζονται αυτές οι δύο ψηφοφορίες. Χωριστά για την ε, συμφωνία της διαπραγματευτικής ομάδας και άλλο ένα πλήν Το κείμενο της Κομισιόν και έχουμε και το παράρτημα της ε, διαπραγμάτευσης. Έτσι, το οποίο είναι παρακολούθημα των άρθρων. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, λέει η Πρόεδρος. Ε, αντιλαμβάνομαι πως δεν το απαγορεύει το άρθρο 70, το να έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Αλλά δεν είναι, και υποχρεωτικό κιόλα. Οπότε είναι στη διακριτική ευχέρεια της Προέδρου ε, και εγώ κρίνω πως ε, δεν θα έχουμε τώρα χωριστή ψηφοφορία. Προτείνω να περάσουμε στην, σε μία ψηφοφορία όπως συμφωνήσαμε με την διαπραγματευτική ομάδα, εκτός εάν οι συγητές ε, θέλουν να πούν κάτι οι διαπραγματευτές. Η πρότασή μου ως πρόεδρο της Επιτροπής είναι αυτή. Οι συνάδελφοι. Αν συνεχίσετε να επιμένετε, ε, δεν, δεν θα έχουμε χωριστή ψηφοφορία και τα σχετικά. Ναι κύριε Ούτζε, να ψηφίσουμε. Πρόεδρε, ζήτησα να μιλήσω για την ημερήσια διάταξη και για διαδικαστικό. Δεν θέλω χωρίς την ψηφοφορία. Ούτε τη ζητώ. Αλλά η πρότασή σας είναι ε, πρόταση. Η, Κομισ... η Επιτροπή μας θα πρέπει να εκφραστεί για τη δική σα πρόταση. Επ' αυτού πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν. Δεύτερον, ζητώ έτσι όπως ψηφίσαμε και στο προηγούμενο θέμα, να ψηφίσουμε και το κείμενο ολόκληρο. Και στη συνέχεια να ψηφίσουμε για το νομοθετικό ψήφισμα και μια τρίτη ψηφοφορία για την ε, διοργανική εντολή. Ακριβώς όπως κάναμε και στο προηγούμενο θέμα. Τουλάχιστον αυτού του είδους την ε, ξεχωριστή ψηφοφορία, σε τρεις ψηφοφορίες δηλαδή, πρέπει να την κάνουμε. Και ας μην κρυβόμαστε, Πρόεδρε, πρόκειται για καθοριστική ψηφοφορία για τα επόμενα 7 χρόνια και για όλα τα θεσμικά όργανα. Γιατί θα δημιουργήσει την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Ή θα το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ε, ή δεν μπορούμε να παριστάνουμε πώ δεν τρέχει κάστανο. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το εξαφανίσουμε το πρόβλημα αυτό με κανονισμούς. Εγώ δεν νομίζω πως ε, θέλουμε να κρύψουμε οτιδήποτε, ούτε να εξαφανίσουμε τίποτα. Απλώς να σας μιλήσω, να σας πω ότι το παγιωμένο κείμενο και το ψήφισμα το ψηφίσαμε τον Ιούλιο. Δεν θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία λοιπόν. Δεν θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Νομίζω πως τελείωσε η συζήτηση, ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Everybody Ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας, 27 υπέρ. Σαφής πλειοψηφία. Έχουμε 3-4 κατά και 10 αποχές, οπότε ε, εγκρίνεται. Από ό,τι κατάλαβα κάποιοι ε, συνάδελφοι θέλουν την ευκαιρία να κάνουν επεξηγηματικές <coughs> ε, δηλώσεις. Επεξηγήσεις ψήφου. Σας δίνω το λόγο λοιπόν, Κωνσταντσε. Επειδή δεν μίλησα προηγουμένως, επειδή ήθελα να εξοικονομήσω χρόνο, όχι, δεν, ε, δεν μίλησες πολύ, Λάμπερτ. Κοιτάξτε, ναι, ναι, με άλλες συζητήσεις, αλλά τώρα νομίζω ψηφίζουμε για μια συμβιβαστική την οποία όλοι μπορούμε να στηρίξουμε και όλες οι πολιτικές ομάδες μπορούν να τη στηρίξουν και ελπίζω πως θα βρούμε την, την πλειοψηφία για αυτή τη συμβαστική και στην Ολομέλεια. Σε αυτή τη φάση όμως μετά από το τελευταίο δια... τριμερή στο Στρασβούργο μετά από 7-8 ώρες διαπραγματεύσεων ήθελα απλά να πω ευχαριστώ σε όλους και από πλευράς του Λάμπερτ στη γραμματεία, στους πολιτικούς συμβούλους, στα μέλη που μας ε, ακολουθούν κάθε φορά προσεκτικά στην ε, διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Και ελπίζω ότι στην επόμενη Ολομέλεια θα είναι επιτυχής η ε, ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Η Ερμήνια Ματσόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να δώσω μια επεξήγηση ψήφο για την αποχή στην οποία προέβηνε. Είναι μια ψήφος ε, ευχαριστήρια απέναντι στους ηγητές ε, για τη δουλειά που έκαναν, αλλά είμαι απόλυτα αντίθετη στο αποτέλεσμα το οποίο επετεύθηκε στην θέση που είναι εξαιρετικά σκληρή του Συμβουλίου σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Νομίζω πως το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή δεν έγιναν σεβαστές σε αυτή τη διαπραγμάτευση. όπου τελικά χάσαμε σε όλα τα κομπικά σημεία που είχαμε πετύχει εξαιρετικά θετικά αποτέλεσμα σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Μιλώ για το πλαίσιο της απόδοσης, την μακροαιρεσιμότητα και την αναστολή των πληρωμών. Ε, είναι πολύ σημαντικά θέματα όπου κάναμε πίσω και όχι μπροστά σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Και να προσθέσω τελευταίο ότι μόλις πριν από ένα μήνα το Κοινοβούλιο ψήφισε μια επιτροπή αυτής της Επιτροπής για την οποία ήμουν εγώ εισηγήτρια και που εισήγε την ε, ρήτρα αποκλεισμού της ε, συγχρηματοδότησης από τον διορθωτικό υπολογισμό του ελλείμματος και άρα τουλάχιστον κατά αυτόν τον τρόπο ε, απάλληνε τις αρνητικές επιπτώσεις της μακροαιρεσιμότητας της οικονομικής που εισήχθη με αυτό το πακέτο. Αντίθετα και αυτή τώρα ε, ανατράπηκε διότι η παράγραφος 19 που προσετέθη με την προσπάθεια των εισηγητών ώστε να δώσουμε νόημα στην εργασία της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου είναι εξαιρετικά δύναμη για να εξουδετερώσει τις αρνητικές επιπτώσεις του άρθρου 21. Η θέση μου και η θέση της ταλικής Αντιπροσωπείας είναι αντίθετη και η αποχή μας απλώς δείχνει την ε, εκτίμησή μας για την εργασία που έκαναν οι δύο συνεισηγητές. Να εξηγήσω πως η διαπραγματευτική ομάδα ήταν σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την ρήτρα επενδύσεων, γιατί νομικώς αυτή η ρήτρα δεν ανήκει σε αυτόν τον κανονισμό. Σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο αριθμιστικό πλαίσιο της μακροοικονομικής πολιτικής που αντιμετωπίζει τις διαδικασίες υπερβολικού ε, ελλείμματος, τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και στο διπλό πακέτο στο δεύτερο κανονισμό του Τούπακ που είναι για την εποπτεία τη μακροοικονομική υπάρχει άρθρο που επιτρέπει την ε, λήψη υπόψη του συγκεκριμένου σημείου και ο Επίτροπος Όλη Ρέν στην τελευταία στο Στρασβούργο εξήγησε πως εφαρμόζει αυτή τη δικασία όπου λαμβάνει υπόψη τη χρηματοδότηση για τη χρηματοδότηση της ε, διαρθρωτικής πολιτικής στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και υπάρχει ήδη πρόταση από την Κομισιόν, μια ολόκληρη λογική για το πώς θα το ενσωματώσουν και τι θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε. Και αυτό που πρότεινε ο εισηγητής ήταν ε, ακόμα κατά της βούλησης ε, της Επιτροπής. Το να λέμε ότι κινούμεθα προς τα πίσω σε σύγκριση με τα τι πρότεινε η Κομισιόν δεν είναι δίκαιο. Γιατί η Κομισιόν στήριξε αυτό που εμείς προζητήσαμε. Και αυτό που πρότειναν οι συγητές ελήφθη υπόψη. Και αναφέρεται η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της εθνικής χρηματοδότησης στην πολιτική συνοχή. Το έχουμε αυτό, έχουμε τη βάση ώστε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ακολουθήσει αυτές τις διαδικασίες. Νομικώς δεν μπορούμε όμως να το ενσωματώσουμε αυτό στον κανονισμό. Και το δεύτερο θέμα για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα και θέλω να σας ενημερώσω γιατί σωστά μην το γνωρίζετε, ότι δηλαδή Ήμασταν ε, μοναχικοί καβαλάριδες. Ήμασταν το μόνο θεσμικό όργανο που αγωνιζόταν εδώ και χρόνια κατά της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Ούτε ένα κάτω μέλος στο Συμβούλιο δεν έχει υποστηρίξει ποτέ ε, σε αυτό το θέση. Και η Κομισιόν μέχρι τελευταία στιγμή ήταν κατά οποιοδήποτε αποδυνάμωσης αυτών των κανόνων Οπότε αυτό που πρότειναν οι εισηγητές σε σχέση με τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι, και αυτό που πετύχαμε είναι άνευ προηγουμένου για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για την Επιτροπή, την Περιφερειακή Επιτροπή το να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και να ληφθεί υπόψη γνώμη μας στην τελική πρόταση της Κομισιόν και τη δυνατότητα να έχουμε ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα προτείνει, από τη στιγμή δηλαδή που θα υπάρχει ανάγκη να ε, προχωρήσουμε σε αυτή τη δικασία. Αντίθετα, για μένα είναι τεράστια επιτυχία. Εγώ από την πρώτη μέρα ξέρετε ότι ήμουν κατά και έστειλα επιστολές επί επιστολών ε, και στον Πρόεδρο και στην Κομισιόν κατά της μακροοικονομικής αιρεσιμότητα. και ξεκολουθώ να είμαι κατά. Μα ο μόνος τρόπος, η μόνη πιθανότητα να και να ξεπεράσουμε την αντίθεση των άλλων δύο θεσμικών οργάνων είναι να βρούμε κάποια συμβιβαστική. Και από όσο μπορώ εγώ να κρίνω, είναι ότι ο συμβασμός αυτός είναι ισορροπημένος και ότι προστατεύει πολλά όσον αφορά τους τελικούς αποδέκτες. Τώρα σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Ματσόνη, ίσως να μην το θυμάστε, αλλά και πριν λίγες μήνες πριν από την έκθεσή σας έστειλα επιστολή στον πρόεδρο Σούλτς για τη ρήτρα ε, επενδύσεων και την ε, εξάλληψη της ε, συγχρηματοδότησης από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Δεν έλαβα ποτέ απάντηση, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τα όσα προτείνατε εσείς στην εκθεσή σας ακολουθούσαν ακριβώς την ίδια γραμμή. Οπότε το ότι καταφέραμε να υπάρχει αυτή η αναφορά στον κανονισμό μας νομίζω πως ήταν τελικά επιτυχία των εισηγητών. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβετε και από πού ξεκινήσαμε ποιοι ήταν οι, οι, υποστηρικτές μας και κοιτάξτε τις κυβερνήσεις σας. Είναι απίστευτο οι κυβερνήσεις να είναι τόσο κάθετα αντίθετες. Και είχαμε και στο κοινοβούλιο συναδέλφους όπως ο Μάκρος Πίπελα που δεν ε, το ήθελαν, άλλοι που το ήθελαν όπως η κυρία Ματζόνη και οι περισσότεροι συνάδελφοι κάποιων πολιτικών ομάδων. Φυσικό είναι, έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, απλώς προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή συμβιβαστική λύση και νομίζω πως εν γέννη το καταφέρνουμε. Ο κύριος Σούτζες ήθελε να μιλήσει. Παρακαλώ, επεξηγήσεις ψήφου μόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ήθελα να κάνω μια επεξήγηση ψήφου και το λέω αυτό πολύ νυφάλια, χωρίς καμιά διάθεση διπαράθεσης. Ε, Πριν από λίγο θύμισα τη σημασία αυτής της ψηφοφορίας και απλώς θέλω να αναλάβω σαφώς τη θέση μου όπως το έκανα και σε σχέση με τη διαδικασία. Εδώ εισάγεται η υπόθεση των εισηγητών και του ρόλου αυτών. Εγώ νομίζω πως θα πρέπει να αφήσουμε το πεδίο ως που, της ευθύνης των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών και τους οποίους ευχαριστώ ξεκινώντας από τον συνάδελφο Ιβάρης Κουτουμάνης που έκανε εξαίρετη δουλειά. Όμως, όπως μας μαθαίνει ήδη, η Καθολική Εκκλησία και το δεύτερο, η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού ε, άλλο είναι το λάθος. Αν είναι λάθος ε, που το κάνει κάποιος χωρίς να γνωρίζει τι συμβαίνει, ε, ε, ε, εντάξει, εκεί φυσικά δεν τίθεται το θέμα, αλλά εδώ όταν εν γνώση μας ξέρουμε ότι θα γίνει, εγώ θέλω να γραφτεί στα πρακτικά αυτό γιατί είναι ιστορική στιγμή ε, και τη στιγμή που αυτή η Επιτροπή, από τη στιγμή μάλλον που ελευθερώνει αυτό το φάκελο η Επιτροπή μας, αφήνει το Κοινοβούλιο και στη Διεργανική Συμφωνία κάτι το οποίο θα είναι, έχει θα είναι εκρηκτικό. Το να λέμε ότι στην πολιτική συνοχή η μακροαιρεσιμότητα και άρα το κενό, το πρόβλημα κάποιων κρατών μελών που πρέπει να συνεχίσουν και να γίνουν και αργότερα εμπόδια και μειονεκτήματα, αυτό σημαίνει δημιουργία Ευρώπης δύο ταχυτήτων, όπου θα υπάρχουν αυτοί που έχουν τους λογαριασμούς τους εντάξει και που θα συνεχίζουν να χαίρουν όλων των χρηματοδοτήσεων και εκείνους επειδή έχουν μακροαιρεσιμότητα που δεσμεύουν την ανάπτυξή τους και την οικονομική τους ε, μεγέθυνση δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα. Και ε, μια τελευταία μικρή παρατήρηση. Όλα αυτά θα αντικατοπτριστούν αρνητικά και στο οικονομικό σύστημα και στο σύστημα των επιχειρήσεων. Γιατί αφού οι χώρες ε, δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε προγραμματισμό των δαπανών για τις χώρες με μακροαρισμότητα και ο οικονομικός τους, δημοσιονομικός προγραμματισμός τα επόμενα 7 χρόνια θα ε, επιβαρυνθεί. Γι' αυτό το καταψήφισα και επαναλαμβάνω χωρίς διάθεση για την παράθεση, η νυφάλια, αλλά έχω το καθήκον να αναφέρω αυτή τη θέση που δεν είναι προσωπική και που είναι απόλυτα ε, κέρια. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να εξηγήσω το γιατί ψήφισα όπως ψήφισα. Αφορά βεβαίως κατά κύριο λόγο την μακροοικονομική αιρεσιμότητα και ε, λυπούμε για το ότι δεν επιτρέψατε χωριστή ψηφοφορία από αυτού. Κατόπιν, αλλάζει εδώ πέρα η φιλοσοφία της πολιτικής συνοχής. Μέχρι τώρα ήταν να προσπαθήσει να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα ε, έχουμε εισαγωγή ενός αντιπαραγωγικού στοιχείου. Δηλαδή τιμωρούνται οι περιφέρειες για αυτά τα οποία κάνουν τα κράτη-μέλη και μπαίνει ένας μηχανισμός στον οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ως ε, κοινοβούλιο. Οπότε δεν βλέπω και κάποιον πιθανό συμβιβασμό. Και δεν είναι δυνατόν δηλαδή να τιμωρούνται οι ασθενέστερες ε, περιφέρειες. Λυπούμε πάρα πολύ και ειλικρινά και εγώ προέρχομαι από μία περιφέρεια η οποία κερδίζει από τον γενικό κανονισμό, αλλά δεν μπορώ να το δω εγωιστικά το ζήτημα. Μπορώ να δω τι προέκυψε συνολικά. Αυτή είναι η αποστολή μας εδώ σε αυτή την επιτροπή. Και Κωνσταντσε, άρα θέλετε να πείτε κι εσείς κάτι. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Το άρθρο εδώ πέρα είναι το άρθρο 21 αυτό το οποίο απασχολεί τους περισσότερους. Και δεν μιλήσαμε για τον συμβιβασμό τον οποίο επιτύχαμε, γι' αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια αν μου επιτρέπετε. Δεν συμφωνώ πάντα με τον Μάρκους Πίπερ, αλλά έχει απολύτως δίκιο και ελπίζω να γραφτεί στα πρακτικά όταν λέει πως το άρθρο αυτό 21 δεν θα εφαρμοστεί τα επόμενα 7 χρόνια. Και αυτή είναι επιτυχία της διαπραγματευτικής ομάδας. Γιατί φτιάξαμε ένα άρθρο 21 όπου η μακροοικονομική ερεσιμότητα έχασε ε, όλη την ουσία σχεδόν που είχε. Έχουμε βάλει τόσο πολύ ε, άμμο στα γρανάζια, δεν μπήκε ως όρος η ανεργία που πρέπει να ληφθεί υπόψη, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός ότι δεν μπορεί να υπάρχει διακοπή των ε, πληρωμών όταν μια χώρα είναι σε πολυετή ύφεση. Ότι μπορεί να περικοπεί μόνο στο τέλος της προγραμματικής περίοδου μόνο ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Και οι χώρες οι οποίες έχουν οικονομικές δυσκολίες ε, πρέπει να έχουν προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας κτλ. Όσες τα κάνουν αυτά εξαιρούνται. <coughs> Εντελώς. Δηλαδή, με όλα αυτά, αυτό το οποίο παραμένει είναι κάτι το συμβολικό. Γιατί επέμενε το Συμβούλιο και 28 ή 28 χώρες, ούτε μία δεν είπε θέλουμε... Ε, να μην υπάρχει μακροοικονομική ερεσιμότητα. Αν διαβάσετε ήρεμα τον συμβιβασμό που πετύχαμε και επιμένετε να ρισκάρετε ολόκληρη την πολιτική συνοχής είναι κάτι που πρέπει ο καθένας μετά να το σκεφτεί. Εγώ θεωρώ πως έχουμε μια καλή λύση, ένα καλό συμβιβασμό και πραγματικά θα ήθελα να υπερασπιστώ τη δουλειά που κάνουμε. Ευχαριστώ η Κωνσταντζέ ξέχασε να πει πως ξεφορτωθήκαμε και το όνομα μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Δεν λέγεται έτσι πλέον. Έτσι. το έχουμε υπόψη. Για να εξηγήσω αυτό το οποίο λέει η Κωνσταντζέ, Γιατί υπάρχουν δύο πτυχές. Το ένα είναι πως παλεύαμε στην Επιτροπή μας χρόνια να μπορέσουμε να βρούμε αυτή τη σχέση μεταξύ τη ε, διακυβέρνηση, του συντονισμού τη πολιτική Ευρώπη και τη πολιτική συνοχή, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική τη συνοχή είναι η βασική πολιτική των επίπεδων Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια έχουμε αναπόσπαστα δεμένο και το εξάμεινο. Οπότε έτσι φαίνεται ποιε είναι οι προτεραιότητε τη πολιτική. Και επίση έχουμε και κάποια θέματα που είναι σημαντικά για ε, τη γενική διδακτική ας πούμε ε, της οικονομικής πολιτικής. Και οπότε και αυτό είχε να κάνει και με τις ε, κυρώσεις, τις θεσπιστήσεις, οπότε και γι' αυτό και η Κωνσταντζα έλεγε ότι όλα αυτά θα πανευρωθούν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω του ε, συνδυασμού αυτών των τριών ε, ε, παραγόντων, παινία, κρίση κλπ. Και όλα αυτά θα οδηγήσουν στην αναστολή ή στο ενδεχόμενο αυτής. Οπότε, δεν έχουν γίνει και λίγα ούτως ώστε να συνδέσουμε αυτές τις μεταβλητές μεταξύ τους. Αυτά τα μέτρα τα οποία να κάνουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων και της ε, οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης. Οπότε τα πράγματα ας μην αλλάξουν και ας ελπίσουμε ότι αυτά θα αξιοποιηθούν, αλλά όπως είπαμε τελικά κανείς δεν είχε δείξει κάποιο που να ανοιχτή στάση, ούτως ώστε να συνομιλήσει με εμά και γι' αυτό και τελικά καταφέραμε κάποιον ε, ε, εύστοχο συμβιβασμό διάφορων στη στο λόγο. Πρώτη, η Ελισάβετ Σουρέντερ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω πως είχαμε συνεργασία με τη διαπραγματευτική ομάδα ε, αρκετά επιτυχή. Καταφέραμε να περάσουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είχαμε το πρόβλημα στην αρχή πως ήμασταν πάρα πολύ ήπιοι. Καταφέραμε να περάσουμε αρκετά σημεία, ακριβώς γιατί ήμασταν ενωμένοι. Και η συνοχή αυτή έσπασε σε ένα σημείο, την μακροοικονομική Η Γεγονός είναι πως προσπαθήσαμε τα πάντα και αυτό το οποίο περιγράφηκε, αλλά δεν προέκυψε ε, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και πράγματι προσπαθήσαμε να το καταστήσουμε τελείως ε, συμβολικό να ξεπεράσουμε το μπλοκάρισμα του Συμβουλίου και να μην ε, μπορέσει να χρησιμοποιήσει το μέσο αυτό. Συμφωνήσαμε, αλλά αυτό το οποίο προέκυψε τελικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πολύ ουσιαστικά σημεία. Δηλαδή η πρότασή μας ήταν ε, να μείνει επί της αρχής μόνο στις υποχρεώσεις και όχι στις πληρωμές. Αλλά, δεν τα καταφέραμε να το περάσουμε αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό το να μην ήταν οι πληρωμές που τελικά είναι μέσα γιατί οι τράπεζες δίνουν πιστώσεις ε, αλλά αν ξέρουν πως δεν θα έχουν την πληρωμή ως εγγύηση στο τέλος γιατί μπορεί να ανασταλούν οι πληρωμές θα είναι πάρα πολύ προσεκτικότερες. Έτσι δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν επιτυχή ε, χρηματοδοτικά μέσα ε, γιατί θα είναι πολύ πιο μαγκωμένες οι τράπεζες. Και κάτι άλλο που από πράσινη πλευρά ξεπέρασε τα όρια την κόκκινη γραμμή. Εξού και η αποχή η δική μας. Γιατί έχουμε ένα ξένο στοιχείο στην πολιτική συνοχής. Για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τη δυνατότητα που ε, έχουμε να γίνει κάτι στην Ολομέλεια και να πάει στη δεύτερη ανάγνωση. Δεν το βρίσκω τόσο κακό αυτό. Τα υπόλοιπα συμφωνήσαμε όλα και εδώ πέρα δεν μετακινήθηκε καθόλου το Συμβούλιο σε αυτό το σημείο. Εάν λοιπόν απορρίψουμε σε αυτά, αν αυτά τα δύο σημεία, το άρθρο 19 και 21 στην Ολομέλεια και το κείμενο της Κομισιόν, τότε θα έχουμε περάσει τη θέση μας, θα υπάρξει μετά δεύτερη ανάγνωση για αυτό το θέμα ακριβώς. Και μόνο με αυτό το θέμα θα επικρατήσουμε νομίζω. Έχουμε δηλαδή τουλάχιστον μια ευκαιρία να το πετύχουμε. Γι' αυτό θεωρώ πως θα ήταν έξυπνο στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε ως εξής, να απορρίψουμε και τη συμβιβαστική πρόταση και το κείμενο της Κομισιόν και να πάμε στην αρχική πρόταση του Κοινοβουλίου, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε μόνο εδώ μέσα, αλλά και στην Ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία. Τότε θα πάμε σε δεύτερη ανάγνωση και θα μετακινηθεί το Συμβούλιο. Γιατί είναι σαφές πως ε, είναι βασικό αυτό το θέμα για μας. Και, και επί της ουσίας βεβαίως νομίζω θα έχουμε έτσι κάνει κάτι. Έτσι μπορούμε να πάμε σε μια δεύτερη ανάγνωση και νομίζω θα έχουμε τελικά επιτυχή κατάληξη για το κοινοβούλιο. Ο κύριος Χρυσόγυλος και παρακαλώ να είστε λίγο σύντομοι συνάδελφοι. ευχαριστώ. Ε, σίγουρα ακούω τα επιχειρήματα και τα ξέρουμε τα επιχειρήματα ότι μπήκαν τόσα πολλά εμπόδια ώστε στο τέλος δεν εφαρμοστεί. Αλλά όμως φοβάμαι ότι το μήνυμα προς τις κοινωνίες και προς τις περιφέρειες είναι ότι άνοιξε το παράθυρο. Δεν άνοιξε η πόρτα, αλλά άνοιξε το παράθυρο για εφαρμογή της, της μακροοικονομικής ερεσιμότητας Και αυτό είναι κακό γιατί η πολιτική συνοχή στην πραγματικότητα είναι η προσπάθεια να μειώσουμε τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών και να έρουμε τα εμπόδια και τις καταστάσεις που έχουν δημιουργήσει αυτή την ανισότητα και την απόσταση μεταξύ των περιφερειών. Παρόλο ότι θέλουμε πάντα να λειτουργεί ένας δίκαιος συμβασμός, νομίζω ότι δεν ήταν και ως ομάδα και νομίζω και άλλοι ευρωβουλευτές το τονίσανε, ε, πιστεύω ότι στην Ολομέλεια πρέπει να καταθέσουμε τροπολογία για να εξαλειφθούν τα άρθρα 19 και 21. Το πρόβλημα είναι ότι και η ύπαρξη μόνο του όρου θα δημιουργήσει αρνητικές οικονομικές προϋποθέσεις και θα επικρέμεται ως απειλή συνεχώς ότι μπορούν να εφαρμοστούν έστω κάποια στιγμή ε, τα κριτήρια της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Και νομίζω ότι οφείλουμε ως Επιτροπή τουλάχιστον Περιφερειακής Ανάπτυξης να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση και στην Ολομέλεια και θα παρακαλούσε και ευρωβουλευτές από την Επιτροπή να καταθέσουμε ε, πρόταση στην Ολομέλεια όταν θα έρθει για ψηφορία ώστε να απαλληθούν τα άρθρα 19 και 21. Α, ε, ήθελα να κάνω παρεπτόντως και μια πρόταση. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ξεκίνησε μία ακρόαση σε σχέση με τις επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών της Τρόικα στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Θα έλεγα να καλέσουμε να ξεκινήσουμε κι εμείς μία τέτοια διαδικασία στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, να δούμε δηλαδή κατά πόσο αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα έχουν επιπτώσεις στην πολιτική συνοχή και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μια διαδικασία που το Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να ξεκινήσει και η δικιά μας Επιτροπή στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και θα παρακαλούσα η Πρόεδρος να πάρει μια πρωτοβουλία να καλέσουμε και εμείς τους εκπροσώπους της Τρόικα αλλά και πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους των περιφερειών να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς τώρα με την κρίση και τις πολιτικές της Τρόικα ε, σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Thank uh, Mr. Κύριος Κοντουμάνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα. Τους συναδέλφους. Ο καθένας μίλησε τόσες φορές, εγώ θέλω να σας πω, ότι συμμετέσχουν στις διαπραγματεύσεις και ήμουν συντονιστής της ΑΛΔΕ ε, για την Επιτροπή μας και είχα πει ότι και εγώ επιφυλάσσομαι γιατί θεωρώ ότι δεν θέλω όλοι αυτοί που μέσω διαδικτύου μας βλέπουν να θεωρήσουν ότι το μοναδικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο 100% της αιρεσιμότητας που ήταν της μακροοικονομικής Και άρχισε μια ματιά στην ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με το μείο Συνοχής. προβλεπόζουν κάποιες ε, χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί στην Ουγγαρία, ευτυχώς για πολύ λίγο, αλλά αυτό δεν είναι μια καινοτομία. Παρακαλώ, μελετήστε προσεκτικά, κυρίε και κύριοι, την ισχύουσα νομοθεσία. Δεύτερον, ναι. Καταρχήν όλα αυτά τα κάνουμε για την κρίση. Η εξαπλή δέσμη, η διπλή δέσμη ισχύει για τις χώρες της Ευρωζώνης και όσους ε, συμφώνησαν να αναδεχθούν τα μέτρα, αλλά η πρόταση τη Επιτροπή ε, έκανε πιο αυστηρές τις ε, ποινέ. Καλά. Συζητήσαμε ευθύς εξ αρχής και ίσως δεν είναι κάτι το για το δίκαιο, αλλά, αλλά κυρίες και κύριοι, για διαβάστε και το παράρτημα συγκεκριμένα τα άρθρα 19-21. Εκεί λέγεται το συμβασμό. Οπότε, πρόκειται περί συμβασμού και είπαμε ότι σε σχέση με την μακροοικονομική εδεσιμότητα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το Συμβούλιο ε, αυξάνει και Είπαμε ότι ή θα πρέπει το πρόγραμμα να τηρηθεί για το έλλειμμα ή αν δεν τηρηθεί το πρόγραμμα τότε θα επιληθούν κυρώσεις. Και βλέπουμε στην αρχή έχουμε 50% μετά έχουμε 100% όσον αφορά την ανισορροπία για το έλλειμμα κλπ. Οπότε για να στάλησαν οι εκταμιεύσεις προς τα σχετικά κράτη μέλη. Αλλά, αλλά εμείς γιατί λέμε ναι, γιατί πρόκειται περί συμβιβασμού. Και βέβαια δεν λέμε όχι σε όλη την πληρωμή, λέμε 50%. Δεν πάμε στο 0, πάμε στο 50%. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και το απέσπασαν οι εισηγητέ. Δεύτερον, έχει να κάνει αυτό με την ε, ανεργία που έχουμε ε, αυτό το ποσοστό αν ε, είναι 2% έχουμε μείωση, αν είναι 5% μεγαλύτερη μείωση. διαβάστε, διαβάστε τι λέει το παράρτημα. Μέχρι 50% μείωση προβλέπεται δεύτερον. Όλα αυτά έχουν να κάνουμε και με την παινία, ε, την κοινωνική ένταξη. Όλα αυτά τα λέει, τα λέει το κείμενο. Επίσης λέει για τη, διπλή συρρήκνωση του ΑΕΠ. Οπότε ακόμα και αν πάτε τα τελευταία δύο χρόνια. 20, 2019, 2018 κατεβαίνουμε είναι οι χρονιές για τις οποίες πρέπει να εγκριθούν αυτά τα κονδύλια και για φέτος το 2013 επίσης υπάρχει μείωση των κυρώσεων σε περίπτωση που αναδεθούν οι σχετικές συνθήκες. Πρόκειται περί συμβασμού κύριε και κύριοι. Και αν κάποιος θεωρήσει το αντίθετο θα κάνει λάθος. Επίσης, έχω να σας πω ότι όχι μόνο αυτό αποσπάζουμε στις δυο διαπραγματεύσεις, αλλά Αντί για 7% πήγαμε στο 6% που είναι πραγματικά ε, χρήματα τάξιος μεγέθους δισεκατομμύριο που θα καταβληθούν μετά το 2020, προχρηματοδότηση, ετήσιο, ποσοστό της ρυθμός, δεν είναι 0,5, φτάνει μέχρι το 3% για το 2020 αποσπάσαμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Οπότε, γι' αυτό σας λέω. Είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα εργαλεία. Να κάνουμε κάτι για αυτή την κρίση. Εντάξει, με έμεσο τρόπο κάνουμε κάτι. Αλλά ας θυμηθούμε την τελευταία φορά που είχαμε κρίση σε ποιο σημείο φτάσαμε. Κοιτάξτε. Διόρθωσε. Τροποποίησε η Επιτροπή το πρόγραμμα για το υπερβολικό έλλειμμα για Γαλλία, για Ισπανία και άλλες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε πρόγραμμα αυτής εξ αρχής και ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν ε, κάτι για του χρόνου. Όλοι Ρεν το μελέτησε και το ενέκρινε έδωσε αναστολή, αναβολή και στην Ισπανία και στην Γαλλία συμβολικού χαρακτήρα μέτρα επομένω. Αλλά εμεί δώσαμε τη μάχη μέχρι το τελευταίο θρόλεπτο. Και επομένω, γι' αυτό σα λέω, είναι πάρα πολύ σοβαρό ο συμβασμό. Οπότε θα πρέπει και πάλι να ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε του εισηγητέ μα. Mr. Mulțumesc, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρως. Εγώ μπορώ να στηρίξω τις προσπάθειε των διαπραγματευτών. Δεν ξέρω αν υπάρχει απαραίτητη εμπειρία από πλευρά Κομισιόν και Συμβουλίου για να διαπραγματευτούν με το Κοινοβούλιο. Βλέπω πως δεν υπήρχε διάθεση για συμβιβασμό που είναι το νόημα της ε, διαπραγμάτευσης. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε εμεί είναι να χάσουμε, να μην έχουμε κατά νου τις σημαντικές ε, πτυχές. Πρώτα απ' όλα. Ε, δεν συμφωνώ 100% με αυτό το οποίο είπε ο κύριο Σόιγκουτμαν για το τι προκύπτει ως αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις για το ότι δεν έχουμε Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Φοβάμαι ότι αυτό ακριβώς αντιμετωπίζουμε. Η πολιτική συνοχή είναι να επενδύουμε ως δυνατόν περισσότερο για να γίνουμε παγκόσμια δύναμη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε Βραζιλία, Κίνα, Ινδία και άλλες οικονομικές δυνάμεις. Εάν πάμε στις χώρες μας και πούμε διαπραγματευτήκαμε τόσο πολύ καλά και τελικά θα πάρουμε λιγότερα λεφτά, δεν θα υπάρχει καμία συνοχή και οπωσδήποτε δεν θα επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Έχλα τώρα να αναφέρω κάποιες άλλες πτυχές. Συγχρηματοδότηση Βεβαίω δεν ήμουν εκεί στι διαπραγματεύσει, αλλά θα, θα έπρεπε να μπορούμε να πάρουμε κάτι παραπάνω από 1%. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να φέρνει τόσε αντιρρήσει στο Συμβούλιο. Υπάρχει ένα παράδοξο επίση το οποίο πρέπει να γνωρίζει η Επιτροπή, το ότι δηλαδή δεν μπορούμε αφενός να συμφωνούμε στην νομοθετική διαδικασία και μετά όταν μιλάμε για κυρώσεις να έχουμε συμβουλευτικό ρόλο. Ο δομημένος διάλογος όπως λένε. Δεν, δεν κολλάνε αυτά τα πράγματα, κάτι πρέπει να γίνει. Ο μόνος λόγος λοιπόν για τον οποίο υπερψήφισα ήταν πως οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι εις βάρος όλων. Νομίζω πως ήταν καλό να δεχτούμε αυτή τη συμβιβαστική λύση. Ψήντω ότι βεβαίως ε, και από πολιτική σκοπιά καλό είναι. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Έρχονται εκλογές, θα πάμε στις χώρες μας και θα πούμε ναι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεχτήκαμε μικρότερο προϋπολογισμό από ότι το 2007-2013 αλλά όσον αφορά την πολιτική συνοχής ε, δεν ε, καταφέραμε να εισακουστούμε γιατί ε, εμφανίστηκε με πολύ σκληρή θέση το Συμβουλίο. Δεν ξέρω αν μας συμφέρει να πούμε κάτι τέτοιο. Οπότε θα ήθελα να πω πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως ε, το ότι έχει απομείνει στο μέσο αυτό όσον αφορά την πλευρά του δομημένου διαλόγου και το ότι δηλαδή είμαστε συνομοθέτες και πρέπει να ακούγεται η φωνή του Κοινοβουλίου. Και βεβαίως να περάσουμε τροπολογία στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Να σας δώσω άλλη μια εξήγηση. Αντιλαμβάνεστε πως κάποια από τα οικονομικά αυτά ζητήματα επηρεάζουν και τη διαμόρφωση των πληρωμών, των πληρωμών σε ολόκληρη την περίοδο. Εμείς ε, δεν μιλήσαμε για τη διαμόρφωση των πληρωμών και τις πληρωμές του προϋπολογισμού, όπως τις πρότεινε το Συμβούλιο. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα βεβαίως να πάμε κόντρα στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου εκεί όπου μπορούσαμε να μετακινηθούμε, όπως είπε και ο κ. Γκοντμάνης, είναι οι ετήσιες προκαταβολές. Για την αρχική προκαταβολή δεν μπορούσαμε να ε, πάμε να διαστέσει το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. μετά από την ε, ψηφοφορία του Νοεμβρίου για το πολιτισμό σου νοικοπλησίου, ο κ. Madame la Présidente, merci. Μετά το σεβαμε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην ψηφορία. Εγώ δεν είμαι κατά αυτή ε, αυτής της συμφωνίας που επιτεύθηκε. Ε, αλλά τελικά η στάση μου δεν είναι εποχή. Νομίζω ότι θα πρέπει Να δούμε ποια θα είναι τελικά η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Γιατί νομίζω ότι τελικά ήμασταν ε, στο ύψο του ρόλου που πρέπει να έχουμε ω συνομοθέτε. Οπότε άπαξ και εξετάζουμε ε, συνολικά αυτόν τον κανονισμό όλοι μπορούμε να παραδεχθούμε ότι οι πρόοδοι τις οποίες επέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με κάποιες προτάσεις ε, τις οποίες εντάξαμε στις ε, διαπραγματεύσεις δεν ήταν και λίγες και ήταν πάρα πολύ πραγματικές, ουσιαστικές. Βεβαίω υπήρχε και το θέμα αυτό που δικαίως μας απασχολεί όσον αφορά την μακροοικονομική αιρεσιμότητα σήμερα δε. Όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι εμείς δώσαμε μία μάχη μέχρι το τέλος όσον αφορά αυτήν την μακροοικονομική αιρεσιμότητα και δικαίως είχαμε στυλώσει τα πόδια γιατί θεωρούσαμε ότι καυτόν τον τρόπο θα είχαμε απονεύρωση της περιφερειακής πολιτικής. Όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, δεν είναι δυνατόν κανείς να θέλει να επιβάλλει σε κάποιες διαπραγματεύσεις ε, κάτι το οποίο ο συνομιλητής αρνείται. Ε, όσο και αν ε, κάποιες φορές, κάποιες φορές λέμε ότι το Συμβούλιο είναι αδιάλεκτο κλπ. κλπ. Μα και εμείς όμως δείξαμε αδιαλαξία μέχρι τη 12η ώρα, αλλά όμως κάποια στιγμή κάτι ίσχυσε η ωρα αλλα ομως καποια στιγμη κατι η υπευθυνοτητα και αποσπάσαμε ένα συμβασμό. Ε, επίσης δε, σε σχέση με την αδιαλαξία του Συμβουλίου, ε, νομίζω ότι καταφέραμε να ε, περιοριστούμε σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία αυτής της ρεσιμότητας. Και αυτό πετύχαμε, δεν είναι ασήμαντα όλα αυτά. Ε, που υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα ε, ε, μέσα οικονομικής πολιτικής που μας ανησυχούν και θα πρέπει να προσέξουμε τόσο ώστε η πολιτική συνοχής, η πολιτική ελληνικής να μην εκτραπεί, να μην γίνει κάτι άλλο και τελικά να μην μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο. Προσωπικά προβληματιζόμαι πάρα πολύ βαθιά σε σχέση με το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής πέραν του 2020. Γιατί έχουμε κάποια ολιστήματα, αυτά τα οποία τώρα εκτιλήσουν. Επίσης τελευταίο να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων της ομάδας διαπραγμάτευσης. Γιατί βοήθησαν πάρα πολύ την απότερη περιφέρεια της Ένωσης και τα σχετικά μας ε, αιτήματα καλύφθηκαν. Και γι' αυτό και θεωρούμε ότι είχαμε σημαντικά βήματα πρώτον. Ναι, βεβαίως, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι αρνητικό το που κατέληξε η υπόθεση της αιρεσιμότητας και ο καθεθένας από εμά μπορεί όλα αυτά να τα διατρανώσει στην Ολομέλεια, όμως από την άλλη μεριά είναι αλήθεια ότι ο γενικότερος συμβασμός ο οποίος κλείστηκε κατά τη γνώμη μου είναι λογικός και επίσης μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη και τον παρόντα χρόνο μια που οι περιφέρειες και αυτές περιμένουν να υπάρξει απέμπλοκη ούτως ώστε αρχές του 2014 να έχουμε ε, τη, το, να αρχίσουν να τρέχουν όλες τις σχετικές διαδικασίες. Βίκτορ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω για κάτι το διαφορετικό. Όπως σας να γνωρίζετε, η διαπραγματευτική ομάδα απέτυχε για δεύτερη φορά να επιτύχει συμβαστική λύση με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για αυτήν την περίφημη κανόνα εν συντρία. Διακόπτη πρόεδρο. Ελπίζω να μην θες να μιλήσει για το δικό σου θέμα, γιατί θα το συζητήσουμε μετά. Για την επεξήγηση ψήφου, ναι. Εγώ θα μιλήσω στη γλώσσα μου, τη μετρική. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να εξηγήσω εγώ πώς ψήφισα. Εγώ υποστήριξα το ψήφισμα, την πρόταση αυτή και συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις και εκεί πέρα βέβαια αντιλήφθηκα πως ο καθένας πρέπει να συμβιβάζεται σε κάποια πράγματα και προσπάθησα να καταλάβω και το τι ήθελε η Κομισιόν. Ήθελε να περάσει κάποιες μεταρρυθμίσεις, να ασκήσει πίεση κτλ. Εγώ ευθύς εξ αρχής ήμουν κατά της ε, μακροοικονομικής ε, αιρεσιμότητας, αλλά ε, η τελική λύση είναι ένα συμβασμός που, που δεν νομίζω πως πρέπει να μας κάνει να ντρεπόμαστε. Αναφέρθηκε ήδη πως λαμβάνεται υπόψη η φτώχεια, η ανεργία, η ύφεση. Υπάρχει κομμάτι για την απασχόληση των νέων κτλ όλα αυτά έχουν μπει μέσα. <clears throat> Πρέπει να το δούμε λοιπόν ως μία συνεισφορά στον διάλογο και καλό θα ήταν να γίνει κάτι ανάλογο και στους υπόλοιπους ε, τριμερείς διαλόγους όπου δεν έχει υπάρξει τέτοια αναβολή. Ε, δεχόμαστε μεγάλη πίεση αλλά ε, σε αυτό θα αναφερθώ άλλη φορά. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα πραγματικά να επενέσω τη διαπραγματευτική ομάδα. Ευχαριστώ Λαμπέρ. Ευχαριστώ για την στήριξη και για το γεγονός ότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από την 1η Ιανουαρίου. Το σημαντικότερο νομίζω σε καιρού κρίσης είναι να διατηρηθεί ο ρυθμός που απαιτείται για να επιφέρουμε τις απαραίτητε αλλαγές στο πακέτο. Και θα πρέπει να εστιάσουμε ακριβώς στην ε, μακροοικονομική ρυθμότητα και τι θα γίνει ε, όταν χώρες πραγματικά δεν ε, μπορούν να ε, ανταποκριθούν σε αυτήν. Είναι πραγματικά το πάρα πολύ δύσκολο. Και, όπως είπαν ήδη κάποιοι, Ήταν ένα ζήτημα ε, στο οποίο καταφέραμε να αποσπάσουμε ε, παραχωρήσεις για να έχει κάποια συναπόφαση για κάποιο ρόλο το, το Κοινοβούλιο. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται όσον αφορά την προληπτική φάση και το πώς, ε, το χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. ο διάλογος μεταξύ Κομισιών, Συμβουλίου και των ειδικών στις χώρες για τις ε, ειδικέ συστάσεις αναχώρα. Πράγματι, είναι ένας διάλογος και μπορούμε να συνεισφέρουμε μιλώντας για το μεγαλύτερο επενδυτικό ταμείο που ε, έχουμε που είναι 45% του προϋπολογισμού επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οπότε... Έχουμε τελικά, όπως είπαμε, αυτή την διορθωτική ε, πτυχή συν τέσσερις συμφωνίες οι οποίες δεν τονίζονται αρκετά. Δηλαδή, ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ ε, σημαντικότερος από αυτά το οποίο είχαμε στο Six Pack και στο Two Pack. Δηλαδή άμα το διαβάσετε και το δείτε, έρχεται η Κομισιόν εδώ πέρα πριν λάβει απόφαση, βλέπουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση, ξεκινάει ένας διάλογος, φέρνουν μια πρόταση, έρχονται εδώ πέρα, δίνουν λόγο. Εντάξει ότι δεν θα έχουμε ε, συναπόφαση πλήρη, ήταν ξεκάθαρο. Αλλά είπαμε. Εξετάζουμε ένα χώρα, το τι γίνεται, την ύφεση κτλ. Οπότε το πακέτο αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε υπ' αυτές τις, ε, τις συνθήκες. Έτσι και δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελε και το, και το Συμβούλιο. Έτσι, καμία χώρα δεν ήθελε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ένα αποτέλεσμα νομίζω της διαπραγματεύσεις που κάνουμε. Ε, δείτε, ε, δούμε και την οικονομική πτυχή οπωσδήποτε, αλλά νομίζω κατάφερε αρκετά και το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία θα, θα ληφθούν υπόψη. Οπότε, αν το δούμε συνολικά, η συνοχή που υπάρχει στην Ευρώπη δεν, δεν χάνεται. Είναι διαφορετική βεβαίως γιατί έχουμε και την εδαφική διάσταση του μπήκε. Είχε ήδη μπει τώρα πλέον εφαρμόζεται, οπότε... μέσω της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και των συνδέσεων της κοινή ε, ανάπτυξης θα οδηγήσει σε μια επιτάχυνση την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα μεταρρυθμιστικό πακέτο, έτσι. Και στο όλο το εύρος του κανονισμού, αλλά και σε σχέση με τις σημερινές ε, προτάσεις. Και μην ξεχνάμε πως είχαμε κάποια ε, κείμενα στα οποία δεν είχε καθόλου διάθεση το Συμβούλιο να κάνει κάτι. Δεν ε, συναντηθήκαμε άδικα 80 φορές με το Συμβούλιο. Προσπαθούσαμε πραγματικά να α, τους κάνουμε να διαβούν το, το Ρουβίκονα. Και δεν νομίζω πως έχουμε εδώ πέρα συνολικά μια οπισθοδρόμηση της ε, συνοχής. Είναι θα έλεγα ένας εξυγχρονισμός της, ένα εξυγχρονισμός της σε μια εποχή ε, στην οποία παραδείγματος χάρη από την Πορτογαλία φεύγουν ε, οι καλά εκπαιδευμένοι άνθρωποι, οι μηχανικοί κτλ. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και προσπαθούμε ακριβώς να προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτές τις δουλειές, αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Δείτε την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχει 60% ε, περισσότερους αυτοκινητόδρομους κατά κεφαλήν από τη Γερμανία. Έτσι. Και κάθε μήνα βγαίνουν 10.000 νέοι απόφοιτοι από τα πανεπιστήμια. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σύνδεση της εκπαίδευσης με, τη, με την κοινωνία, με το πρασίνισμα που το το βάζουμε μέσα. Όλα αυτά σε ένα νέο πακέτο όπου πραγματικά λέμε πως ε, θα, πάνε, θα πάει ένα 50% σε, αυτό το, σε αυτής μορφής της επενδύσεις. Για να έχουν τη δυνατότητα, όπως είπα, οι άνθρωποι να δουλεύουν στο στο αντικείμενο και τις, τις τους, τους, ε, είτε είναι βιολογικές επιστήμες, ε, ε, αυτοκινητοβιομηχανία, οτιδήποτε. Και βεβαίως να υπάρχει πολύ καλύτερη συνεργασία στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι δυνατότητες τις οποίες δίνουμε κίνητρα αυτή τη στιγμή. Αύριο οι δύο επίτροποι, ο κύριος Χάν ε, και η κυρία Γκίγεν Κουίν, έρευνας ε, δηλαδή και περιφερειακής ανάπτυξης, μαζί με τις ε, περιφερειές, θα αρχίσουν να δουν, όπως είπα, αυτό το θέμα της, την έξυπνη εξειδίκευση. Σύντομα θα έχουμε εδώ πέρα και τα Εθνικά Κοινοβούλια να συζητήσουμε το τι θα περιέχει αυτό το πακέτο και πολλοί έχουν την ιδέα πως η πολιτική αυτή ήταν αυτή η οποία ήταν πριν από 10 χρόνια. Είναι λοιπόν τώρα μια συνοχή η οποία εστιάζει πάρα πολύ περισσότερο στην αηφορία, στις δουλειές και το τι χρειάζεται στις περιφέρειες που δεν είναι μόνο υποδομές. Δεν εστιάζουμε μόνο σε μία πτυχή και λέμε αυτή είναι η πολιτική ε, κατά της κρίσης. Πρέπει να καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για να διατηρηθεί η οικονομική ευρωστία της Ευρώπης και αυτό πρέπει να γίνει τώρα και νομίζω και οι υπόλοιπες ομάδες πρέπει να αναρωτηθούν το εάν εντάξει και εγώ μπορεί να μην είμαι πλήρως ικανοποιημένος αλλά να δούμε εάν θα μείνουμε μόνο στην ε, μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Αν δούμε ή αν θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα πακέτα που έχουν συμφωνηθεί. Πράγματι θα έρθουν και τροπολογίες, αυτό είναι σαφές, το ξέρουμε. Και, και για την Ελλάδα. Παραδείγματο χάρη και η Ελλάδα πρέπει να το σκεφτεί αυτό. Νομίζω έχει με τη νέα προσέγγιση πολύ περισσότερες δυνατότητες από το να επενδύει δισεκατομμύρια σε αυτοκινητόδρομους και νέα αεροδρόμια. Έτσι. Και μετά από... ή να χτίζουν και άλλες χώρες. Χτίζουν αεροδρόμια και σε δύο-τρία χρόνια κλείνουν τα αεροδρόμια και χρεοκοπούν. Έτσι. Οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να διακρίνουμε το, την μεταρρύθμιση που έχουμε επιφέρει και την μία, την μία αυτή πτυχή της ε, μακροοικονομικής αρισιμότητας. Εγώ έτσι τα βλέπω. Σας ευχαριστώ Νίκο, μισό λεπτάκι. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, πράγματι, ε, θέλουμε μια συνεκτική πολιτική συνοχή και σε ορισμένα πράγματα που στον ο συνάδελφο κύριο Νιστερό ή συμφωνώ. Νίστερο, συμφωνώ. Αλλά κοιτάξτε, μερικά παραδείγματα. Η Ελλάδα πράγματι συνεχίζει να επιμένει στο να κάνει του τέσσερι μεγάλου αυτοκινητοδρόμου. Παρόλο ότι ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θεωρεί ότι μόνο οι δυόμιση είναι βιώσιμοι οικονομικά. Αλλά ξέρετε όμω ότι έχουν υπογραφεί οι συμβάσει που αν η Ελλάδα εγκαταλείψει το σχεδιασμό αυτό πρέπει να πληρώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Και εκεί οι εταιρείε είναι γερμανικέ, γαλλικέ και ισπανικέ. Άρα λοιπόν να είμαστε λίγο ειλικρινεί. Δηλαδή πράγματι πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο ανάπτυξη. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει να, παίρνουμε, να παίρνει η χώρα 600 εκατομμύρια από τα προγράμματα περιφερειακή ανάπτυξη για να ενισχύσει τη χρηματοδότηση των αυτοκινητοδρόμων που ξέρουμε δεν είναι βιώσιμη. Δηλαδή πληρώνονται προκαταβολικά πριν καν έχουν φτιαχτεί. Εκεί πρέπει να παρεύουμε όμω, λέω, ω και Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη και να καλέσουμε εδώ τι περιφέρειε να μιλήσουμε για αυτά τα προβλήματα. Να δούμε. Και στα θέματα τη ανεργία. Δεν υπάρχουν χρήματα για να ξεκινήσει κάποιο σήμερα μια κοινωνική επιχείρηση ή να ξεκινήσουν νέοι άνθρωποι επαγγέλματα. Δεν μπορούν να βρουν από το συστημικό τραπεζικό σύστημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα γιατί πρέπει να βάλουν εγγυήσει στα σπίτια του ή κάτι άλλο ακίνητη περιουσία και από την άλλη μεριά δεν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης. Αν δεν υπάρξει λοιπόν μια συνεχτική πολιτική, προφανώς δεν θα πετύχουμε ούτε του δημοσιονομικού στόχου. Γιατί αυτή τη στιγμή το χρέος από 109% έχει πάει πάνω από 168% παρότι έγινε το κούρεμα με το PSI Plus ύψου 107 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή αντί να μειωθεί το χρέος με όλα τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής έχει εκτιναχθεί σε μη βιώσιμα επίπεδα ακόμα και αν γίνει και άλλο κούρεμα, πάλι δεν θα είναι βιώσιμο. Δηλαδή θα είναι στο 120%. 122%. Είναι βιώσιμο αυτό σε μια χώρα που πρέπει να πετυχαίνει 5% πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι αδύνατο. Ποια χώρα πετυχαίνει σήμερα στην εποχή της κρίσης 5% πρωτογενές πλεόνασμα να μπορεί να αποζημιώνει. Επομένως, πρέπει να δούμε τι σημαίνει δημοσιονομική, μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Γιατί προφανώς, ναι, πρέπει να, να υπάρξει εξορθολογισμός των δημοσιονομικών. Our policy... Now, the, the policy changes that we Yes, yes, of course. Από αυτούς και η ομάδα η δικιά μας είναι από αυτούς που θέλουν αλλαγέ, γιατί δεν ήταν βιώσιμο το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Δεν ήταν βιώσιμα τα οικονομικά της. Πρέπει να γίνουν όμως με ένα δίκαιο, ορθολογικό τρόπο, κοινωνικά ισόρροπο. Ξέρετε ποιο είναι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα όλη αυτή τη δημοσιονομική προσαρμογή. Ότι έχει καταστραφεί πλήρω η παραγωγική βάση, έχουν κλείσει 100.000 μικρομεσαίε επιχειρήσει, έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργου, σχεδόν ένα στου τρει μικρομεσαίου πλέον δεν μπορεί να πληρώσει ασφαλιστικέ φορέ και έχουμε 3 εκατομμύρια ανασφάλιστου. Το 30% είναι ανασφάλιστοι, δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγεία. Πώ θα πετύχουμε δημοσιονομική προσαρμογή. Θέλω να ολοκληρώσω τη συζήτηση και να πω να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συμμετείχαν στη συζήτηση και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους. Όλοι μας έχουμε ανησυχίες, αλλά πιστεύω πως σήμερα στόχος είναι να ε, το έχουμε φτιάξει μέχρι τον Ιανουάριο και να κρίνουμε το σύνολο του κανονισμού. Νομίζω πως ως Κοινοβούλιο έχουμε εισάγει πάρα πολλές αλλαγές που θα βελτιώσουν την πολιτική και τις δυνατότητές της να δώσει ε, θέσεις απασχόλησης, ε, δουλειά κτλ. Να ευχαριστήσω τους συζητητές και όλη τη διαπραγματευτική ομάδα γιατί έκαναν εξαιρετική δουλειά όλοι οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ ως Πρόεδρος γι' αυτό. Α, συγγνώμη, δεν σας είδα. Ε, ε είναι και ουσιαστικό και διαδικασία θέμα. Ε, στην πρόταση που έκανε και στη δευτερολογία του κυρίου Χρυσόγελου. Ε, νομίζω ότι ο κύριος Χρυσόγελος αναφέρθηκε περισσότερο ότι η κάθε μας παρέμβαση για την πολιτική συνοχή πρέπει να συσχετιστεί με τις πραγματικές συνθήκες που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη και κυρίως στις χώρες συνοχής. Και ανέφερε το παράδειγμα της χώρας μας, υποστηρίζοντας ε, την ανάγκη να δει και η Επιτροπή μας την αξιολόγηση των πολιτικών σε έκτακτες συνθήκες και με έκτακτα μέσα έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα δώσει πολλές ιδέες για την παρακολούθηση που μπορεί να έχει η Επιτροπή μας στις χώρες συνοχής που είναι κυρίως σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ξεχωρίσουμε από τον κανονισμό που ψηφίζουμε σήμερα διότι η παρακολούθηση της κατάστασης και της πολιτικής συνοχής στις χώρες με προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής δεν έχει σχέση μόνο με ένα καλό πακέτο, έχει σχέση με μια ευρύτερη πολιτική. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Εγώ υποστηρίζω τη συμφωνία και υποστηρίζω και την πρόταση του κυρίου Χρυσόγελου για να γίνει αυτή η ακρόαση στην Επιτροπή μας. Αλλά το λέω για τους συνοδέλφους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα προβλήματα αυτά της Τρόικας και το, ε, της πολιτικής των προγραμμάτων προσαρμογής ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να τα αλλάξουν απόψεις οι συντονιστές για την πρότασή σας. Εδώ θέλω να ολοκληρώσουμε και πάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Μπορείτε να μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα για τον κανονισμό αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Το είπα, το είπαμε. Ό,τι λαμβάνεται υπόψη είναι οι δυσκολίες ε, των κρατών μελών. Το πρώτο κομμάτι αφορά την ε, άρση, όπως είπα, της ε, δέσμευσης των ε, κονδυλίων. Δηλαδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακριβώς τις ε, χώρες ε, που το χρειάζονται περισσότερο. Το δεύτερο κομμάτι αφορά μία επιπλέον αύξηση της συγχρηματοδότησης κατά 10% και παράταση των προθεσμιών και επιπλέον ε, μεταφορά μεταξύ των ε, αξώνων ε, προτεραιότητας. Επίσης πρέπει να πω πως εμείς ήμασταν διατεθειμένοι και για περισσότερη ευελιξία πέρα από την πρόταση δηλαδή της Κομισιόν και του Συμβουλίου στην περίπτωση στην οποία, όπως είπα, είχαμε συμφωνία για την επιπλέον συγχρηματοδότηση. Είχαμε όμως ε, προβλήματα με το σημείο 78 στον πρώτο τριμερή διάλογο τον Οκτώβριο. Ε, υποσχέθηκε η Κομισιόν να υποβάλει μια συμβαστική πρόταση γιατί εμείς θέλαμε να αυξήσουμε το ε, την επιπλέον σχερματοδότηση στην ε, Κύπρο, Ρουμανία, Ιρλανδία, Λετωνία κάτι το οποίο βεβαίως ε, θα οδηγούσε και στο ότι δεν θα είχαμε και πλήρη απορρόφηση των κονδύλιων. Είχαμε ακόμα 2,3 δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, αλλά η Κομισιόν ε, δεν είχε διαθέσιμα τα κονδύλια, γι' αυτό ήταν ε, εναντίον. Τελικά, χτες ε, στην Κορεπέρ συζητήθηκε το θέμα και είπαν πως θα μπορούσε να επεκταθεί η συγχρηματοδότηση όσον αφορά την Ουγγαρία μιλάμε για ένα ύψος 500 ε, ε, εκατομμυρίων ε, ευρώ. Πρόταση η οποία όμως δεν υποστηρίχθηκε κατά πλειοψηφία και χτες το απόγευμα στον τριμερή διάλογο επίσης δεν καταλήξαμε σε κάποια συμφωνία. Επέμειναν στην πρόταση του Συμβουλίου. Έτσι απίθυνα έκλεισε εγώ στα άλλα δύο θεσμικά όργανα και είπα πως δεν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση ε, όταν μιλάμε για διαπραγματεύσεις ε, ισότιμων ε, εταίρων. Δεν ζητάμε. Εμείς, εμείς ζητάμε μια νέα πρόταση με διαφορετικό προπολογισμό. Τώρα αναζητήσαμε κάποια άλλη λύση, δηλαδή να μειωθούν τα ε, ανώτατα όρια και να μοιραστούν οι πληρωμές ε, σε σειρά ετών. Δηλαδή υπάρχει κάποιο περιθώριο. Οπότε ο χτεσινός διάλογος ε, τερματίστηκε, ως, τερματίστηκε έτσι και θα συνεχιστεί την τρίτη του Στρασβούργου και ελπίζω να το συζητήσουμε το θέμα στην συνεδρίαση και να ψηφίσουμε στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου της Επιτροπής μας και τον Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Αυτά όσον αφορά τις χτεσινές εξελίξεις. Μάλιστα, πριν δώσω τον λόγο στον Βίκτορα Μποστινάρο, να πω πως η πρόκληση είναι πως πρέπει να, πρέπει να ψηφιστεί αυτό και να τεθεί ενισχύ φέτος, έτσι. Γιατί εκπνέει ο κανονισμός που έχουμε τώρα. Βίκτορα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να μιλήσω εν συντομία στα ρωμανικά. Ε, καταρχήν να συγχαρώ την Κωνσταντζή και τον Λάμπερχτ για το αξιοσημείωτο αποτέλεσμα που επέτυχαν και το οποίο εγκρίναμε σήμερα εδώ. Γιατί οι κυβερνήσεις μας πραγματικά μας κρέμασαν. Τώρα, για το 1 συν 3 και τα σχόλια του εισηγητή κύριε, κύριο Οι δύο τριμερείς απέτυχαν. Οι δύο απέτυχαν στο να βρουν συμβιβασμό. Αυτό λοιπόν το ξέρουμε και έχουμε και μία ε, φοβερή ανάγκη να ολοκληρώσουμε αυτές τις συζητήσεις γιατί ο χρόνος είναι εις βάρος μας που περνάει. Έχοντας το αυτό υπόψη, ε, να πούμε ότι Αυτές, ε, αυτό συνέβαινε για όλους μας εκείνη την ε, ημέρα. Οπότε κυρία Πρόεδρε σας παρακαλώ δώστε μας ένα χρονοδιάγραμμα επίγων, επίγουσας κατάστασης για να δούμε πόσα θα τα βγάλουμε πέρα. Αυτό που επίσης θέλω να πω είναι ότι θα γίνει η νέα συνεδρίαση εδώ στις Βρυξέλλες και τα προβλήματα αυτά θα συζητηθούν εκεί. Και μια συμβιβαστική θα μπορούσε να είναι αυτή ε, πάντως σίγουρα θα γίνει αυτή η συνεδρίαση και αυτό επιβεβαιώθηκε από το Συμβούλιο και από την ε, Κομισιόν. Την Τετάρτη το απόγευμα θα πρότεινα λοιπόν να οργανώσουμε ένα τριμερί που θα λάβει υπόψη τις συμφωνίες που επετέφθησαν στην Κορεπέρ είτε την Τετάρτη απόγευμα είτε την Πέμπτη ανάλογα με το δικό σας χρονοδιάγραμμα και μετά την επόμενη Τρίτη στο Στρασβούργο θα πρότεινα μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας γιατί βέβαια θα είναι όλοι στο Στρασβούργο για να εγκρίνουμε το αποτέλεσμα του επερχόμενου τριλόγου και έτσι ώστε η ψηφοφορία μας να υποβληθεί στην Ολομέλεια και να ψηφιστεί στη διάρκεια της επόμενης συνεδρίας του Στρασβού, Συνόδου του και όχι αργότερα, γιατί και πάλι, όπως είπα, ο χρόνος είναι εναντίον μας. Συνέταξα αυτή την ε, πρόταση σε συνεργασία με το ΕΛΚ, την ΚΟΥΕ και τους Πράσινους. Παρακαλώ λοιπόν να δεχτείτε αυτό το ε, πρόγραμμα γιατί ε, πρέπει να κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση. Οι χρονικοί περιορισμοί για το συγκεκριμένο θέμα είναι μεγάλοι και για τα ενδιαφερόμενα κράτη φυσικά και πρέπει να εξαλείψουμε κάθε είδους ε, κίνδυνο ώστε να μπορέσει να υποβληθεί και να συζητηθεί η έκθεση τον Δεκέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βλάσακ. Eh, Já ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στους ε, συναδέλφους πως γνωρίζω πως ε, ο χρόνος μας πιέζει, αλλά από την άλλη πρέπει να έχουμε <coughs> κατά νου πως το Συμβούλιο δεν ήρθε με κανένα συμβιβασμό στο διάλογο δεν αποτύχαμε εμείς. Δεν ε, υπέβαλε καμία πρόταση διαφορετική. Δεν, δεν προχωράνε έτσι οι διαπραγματεύσεις. Ακούστηκε πως υπάρχουν άλλες ε, πιθανότητες και πως πρέπει να δώσουμε χρόνο στο Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία με μια διαφορετική ε, συμφωνία ε, από αυτά τα οποία, διαφορετική από αυτά τα οποία είπαμε χθε το βράδυ. Εγώ συμφώνησα και με την Προεδρία και με την Κομισιόν πως το καλύτερο θα ήταν να συναντηθούμε τρίτη στο Στρασβούργο και να συμφωνήσουμε και πως αν συμφωνήσουμε δεν υπάρχει πρόβλημα μετά να το συζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα να τηρηθεί η χθεσινή συμφωνία. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα δεν μιλάω ως συγητής, ως συντονιστής του ΕΛΚ. Οι διαπραγματεύσεις ε, έχουν μία δική τους διάσταση. Μία από τις διαστάσεις είναι ο χρόνος είναι ξεκάθαρο πως ο χρόνος είναι τόσο περιορισμένος ώστε θα έπρεπε νομίζω να, να έχουμε τελειώσει προχτές έτσι αλλιώς θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μία άλλη ε, επιπλέον συνεδρίαση της ε, ομάδας μας. Ε, ο κύριος Βλάσσακ λέει πως δεν πρέπει να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα. Εγώ νομίζω πως πρέπει. Πρέπει να... αφήσουμε βεβαίω ε, τους διαπραγματευτές να κάνουν την, ε, τη δουλειά τους, αλλά... Κοιτάξτε, το πώς θα κυλήσουν τώρα οι διαπραγματεύσεις. Ε, εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Οι σοσιαλιστές ε, έχουν μια διαφορετική τακτική <coughs> ίσως, ε, αλλά εμείς είμαστε διατεθειμένοι, όπως είπα, να κάνουμε την επιπλέον προσπάθεια, να το δούμε το τι θα έχει προκύψει στην ε, εβδομάδα του Στρασβούργου και νομίζω το χειρότερο θα είναι η δυνατότητα που θα προσφέρεται τελικά να είναι τόσο άσχημη, αλλά να μην έχουμε καμία άλλη εναλλακτική και να μην μπορούμε να, να κάνουμε τίποτα άλλο στο τέλος. Έτσι. Πρέπει να έχουμε... Συνάδελφοι, παρακαλώ να είσαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Είμαι και να σα ενημερώσω την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι πολύ δύσκολο τα διότι οι σοσιαλιστές λείπουν όλη τη βδομάδα. Εκτό μικροφώνου, κύριε Ζεμπαστινό. Ναι, ναι, και το ΕΛΚ κάποιε μέρε λείπει. Οπότε προσπαθήσαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Οπότε, οπότε μπορούμε την Τρίτη του Στρασβούρου κάτι να κανονίσουμε. Μετά τι άλλο έχουμε, την Τετάρτη, η μόνη ευκαιρία για να κάνουμε την έκτακτη συνεδρίαση ε, πρωί, αλλά τότε δεν έχουμε χρόνο για τις τροπολογίες. Άρα, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι δυνατόν να προφτάσουμε να ψηφίσουμε μέχρι και την ε, σύνοδο του Νοεμβρίου. Συνεχίζουμε να διερευνούμε τι μπορεί να γίνει, αλλά τα πράγματα είναι πολύ στριμωγμένα. Κωνσταντς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρω με αυτό το οποίο είπε ο Βίκτορ. Εάν υπάρχει κάποιος τρόπος τρίτη του Στρασβούργου το πρωί να κάνουμε κάτι και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε τριμερή διάλογο. Εγώ μπορώ να πω πως ε, εντάξει εμείς έχουμε συνεδρίαση της ομάδας μας αλλά οι αρμόδιοι για την διαπραγμάτευση αυτή θα είναι παρόντες ε, ε, αν είναι να οργανωθεί ένας τριμερής διάλογος και μια που ξέρω πως είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να έχουμε ένα, ένα περιθώριο παραπάνω. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις 14 ε, μέρες του Δεκεμβρίου. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε με, τον, ε, με το Συμβουλίο. Αν το αναβάλουμε κατευθείαν για Δεκέμβριο είναι πλέον τελευταία ευκαιρία και τελείωσε. Μετά θα μπορούμε να διορθώσουμε τίποτα. Έτσι. Μετά αυτό είναι και τέλος. Οπότε θα ήθελα να προσπαθήσουμε να προσπαθήσουμε πράγματι να το κάνουμε την, την επόμενη εβδομάδα. Και, και να έχουμε και μία συνεδρίαση επιπλέον της ομάδας. Ναι, ναι, ε, να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για να έχουμε την ψηφοφορία τον Νοέμβριο. Θα το τσεκάρουμε, αλλά όπως είπατε δεν, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Κύριε Λούχαν, είναι, είναι πολλοί ομιλητές και έχουν μείνει 10 λεπτά. Παρακαλώ λοιπόν. Κυρία Πρόεδρε, οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει ο τριμερής διάλογος πριν την κορεπέρ της Πρέσβης. εβδομάδας. Τέλος πάντων, όσο γίνεται συντομότερα, κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Βλάσεκ. Ήταν κάπως η τοπαθή, η παθητική στάση σε αυτό το οποίο έλεγε αν όλα πάνε καλά, καλώ, αν όχι πάλι πήρα, αλλά εμεί ω Περιφερειακή Επιτροπή θα πρέπει να έχουμε άλλου είδου τοποθέτηση. Συμφωνώ με την Κωνσταντζα, συμφωνώ με τον Λάμπερτ, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να αποσπάσουμε κάποια ε, συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και να δούμε γιατί δεν τα καταφέραμε το βράδυ. Ε, ξέρουμε γιατί προσπάθησε κάτι να κάνει ο σκιώδης ηγητής, αλλά κυρίως για τη χώρα του. Παρά το ότι το Συμβούλιο είπε ότι αυτά όλα θα γίνουν αλλιώς και όχι όπως ήθελε εκείνος. Ήθελε να προωθήσει τις θέσεις του ΕΛΚ και είπε εγώ αυτό θέλω, αυτό θέλω να γίνει παρά το ότι εδώ πρόκειται περί συμβασμού, πρόκειται περί τριμέρους διαλόγου. Τέλος πάντων θα πρέπει να επιδειχθεί ο πολιτική. Να εξασφαλίσουμε το ότι θα εγκριθεί τελικά αυτή η έκθεση. Μήπως ο Δεκέμβριος είναι πολύ αργά. Για να κάτσουμε να δούμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε το πώς όλες οι θέσεις θα συγκεραστούν. Έχουμε, λέει πρόεδρο, την κατάσταση του Συμβουλίου. Η κατάσταση εκεί πέρα είναι ένα διέξοδο με τη Λιθουανία κλπ. Και θα πρέπει όμω να συμφωνήσουν πολιτικέ ομάδε πριν πάμε στον τριμερή διάλογο. Κύριε Μαρινέσκο, ευχαριστώ πρόεδρε. Οπότε έγινε αυτή η προπαρασκευαστική συνάντηση του ΕΛΚ και τα είπαμε και θα κάνουμε την τριμέρη συνάντηση την επόμενη εβδομάδα και όπως είπε ο κ. Βλάσεκ, έτσι είναι. Θα πρέπει κάτι να προκύψει από το Συμβούλιο, αλλά ε, η συνάντηση είναι Τετάρτη το πρωί η συνάντηση του Συμβουλίου. Άρα θα έχει την ίδια θέση το Συμβουλίο. Είτε τα απόγευμα τα πούνε, είτε την Τρίτη, είτε το πρωί. Ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι εάν γίνει ο τριμερής διάλογος Τετάρτη το απόγευμα, υπάρχει κάποια ελπίδα συμφωνίας. Και άρα την πέμπτη στη διάσκεψη των Προέδρων η έκθεση θα μπει στην ημέρησια διάταξη και θα ψηφιστεί στη Σύνοδο. Οπότε και στην έκτακτη συναντήσή μας θα ψηφίσουμε τρίτη πρωί, τετάρτη, πέμπτη, θα ψηφίσουμε ή στην Ολομέλεια. αυτή είναι η διαφορά. Και εγώ ταπεινά σας ζητώ, Πρόεδρε, να ακολουθήσετε αυτή τη μέθοδο, αυτό το τρόπο. Γιατί αλλιώς το Δεκέμβριο, αν πάμε, ε, τότε θα έχουμε πολλές πιθανότητες να μην προφτάσουμε τη δημοσίευση στην επίσημη, στο επίσημο δελτίο και άρα τίποτα, για όλοι θα χάσουν ναι, ναι, ναι, το, το, ζητείτε αυτό, αλλά χθε συμφωνήσατε στον ε, διάλογο να μην γίνει διάλογο, να μην γίνει τριμερή διάλογο την επόμενη εβδομάδα. Τώρα όμω. Μπουστινάρου. Για ενημέρωσή σα. Κομισιόν και Συμβούλιο λένε ότι μετά την κορεπέρα να πάσα στιγμή είναι έτοιμοι να ε, συναντηθούν μαζί μα. Καλά, σύλλα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. ρισκάρουμε την απώλεια 5 δις. Διότι από αλληλεγγύη με τους συναδέλφους χτες δεχθήκαμε συνεχή συζήτηση και μιλάμε για 500 εκατομμύρια από την μια πλευρά αλλά από την άλλη ρισκάρουμε 4 δις. Ναι, λέγαμε. από αλληλεγγύη να πάρουν αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια, αλλά μην χάσουμε τα δις. ε, μιλάμε διαδικαστικά, λέει ο κύριος ε, αλλά ο κύριος Γκουτμάνης, ε, έχουμε τη Σλοβακία και τη Ρουμανία και είναι τα θέματα με τις πιστώσεις υποχρεώσεων και οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια παράταση εκεί της δυνατότητας εκταμίευσης και η Σλοβακία είναι 7η στη λίστα, υπάρχουν χώρες σε πολύ χειρότερη κατάσταση, όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε έβδομη κατάσταση. Θα πρέπει κάτι να γίνει. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε τουλάχιστον για αυτές τις δύο χώρες, διότι εάν δεν συμφωνήσουμε για τίποτα, ε, τελικά και αυτές οι δύο χώρες θα μείνουν ξεκρέμαστες. Αυτό να παρατεινεται si αυτη η κατασταση θα πρεπει κατι να γινει θα πρεπει να συμφωνησουμε τουλαχιστον για αυτες τις δυο χωρες διοτι εαν δεν συμφωνησουμε για τιποτα τελικα και αυτες οι δυο χωρες θα μεινουν ξεκρεμαστες αυτο να καταλαβουμε Όντω μπορεί να δώσει τη μάχη του, αλλά πάντοτε θα πρέπει να ξέρει πού να σταματάει. Αλλιώ. θα πρέπει να δούμε μην μείνουμε στο τέλος με άδεια χέρια. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ με τα συμφέροντα που υποστηρίζει ο εισηγητής στον τριμερή διάλογο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αφήσουμε να χαθούν όλα, να χαθούν και αυτά δηλαδή που έχουμε ήδη επιτύχει. Και γι' αυτό συμφωνώ με την πρόταση του συναδέλφου Μποστινάρο έτσι ώστε να καταφέρουμε να φτιάξουμε σε μια λύση όσο γίνεται πιο κοντινή με αυτή που, μας, που θέλουμε όλοι μας. Ευχαριστώ. Το μήνυμα σας είναι ξεκάθαρο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να είμαστε έτοιμοι πριν από τη διάσκεψη των Προέδρων της Πέμπτης. Μίλησα εχθές με την Προεδρία. Υποσχέθηκαν ότι θα δουλέψουν από αυτού του νέου συμβιβασμού. Ε, κάνουν ό,τι μπορούν και αυτοί δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Να πω στον κύριο Λούχαν ότι τριμερίς πριν από την Κορεπέρ θα ήταν ε, κάτι παράλογο. Δεν μπορεί παρά να γίνει μετά από τη συνεδρίαση του, ε, της Κορεπέρ. Γιατί δεν καταφέραμε κάτι καλύτερο τώρα εχθές. πρόταση της Επιτροπής, δεν, της Προεδρίας με δεν έγινε δεκτή. Ε, δεν προτάθηκε συμβαστική μετά την Κορεπέρ. Ε, δεν υπήρξαν δυνατότητες διαπραγμάτευσης. Εάν φοβάστε πως τα μέσα για την Ρουμανία και τη Σλοβαϊκή θα χαθούν, εάν θέλετε να αποφύγετε την μείωσή τους, λέω εξ αρχής ότι η τελευταία μεταβλητή που έχουμε στην επιτάπη τους είναι αυτή. Αν οι εκπρόσωποι των ομάδων μου πούν πως έχουν μια άλλη άποψη από αυτή που ε, έχει εγκριθεί μέσα στην εντολή, τότε έχουμε πρόβλημα. Χθες ξεκίνησα από μια άλλη οπτική γωνία. Και επιβεβαιώθηκε αυτή μου η άποψη. Προσπαθήσαμε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με την εντολή που είχαμε λάβει. <laughs> Can you do it afterwards, or you have to respond now? Πρέπει τώρα να απαντήσετε, δεν μπορείτε να απαντήσετε μετά. Ο κύριο Βλάσεκ αναφέρθηκε σε αυτά που είπα εγώ πριν προηγουμένως και γι' αυτό θέλω να πάρω το λόγο τώρα. Να θυμίσω στον κύριο Βλάσεκ ότι είναι επικεφαλή των διαπραγματεύσεων, ότι είναι εισηγητής μα και ότι είναι υπεύθυνο για τι διαπραγματεύσει. Ίσως να το ξέχασε το συγκεκριμένο στοιχείο ή να μην του δίνει τόσο μεγάλη σημασία. Όσον αφορά τώρα την χρονισμό των διαπραγματεύσεων θα ήταν πολύ καλά να είχαμε μια θέση εχθές, κύριε Βλάσεκ. Ακόμα κι αν ε, έρχονταν η άλλη πλευρά, ε, με άλλη διαφορετική θέση. Η θέση του κυρίου Τόιτσε δεν είναι η θέση του ΕΛΚ συνολικά. Το είπαμε αυτό και χτες. Η θέση μας είναι διαφορετική κατά τη διάρκεια του τριμερούς. Μπορούμε και αυτό να το αποφασίσουμε επίσης. Μπορούμε να επαναλάβουμε τον χθεσινό τριμερή διάλογο όπου ο κύριος Βλάσεκ ε, ε, ξέφρασε τη θέση του που και όπου όλοι πρέπει να θα χάσουμε αν δεν στηρίξουμε το Συμβουλίο. Μαριάν, να σας πω μόνο πως το πρωί στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση έγινε σαφής πρόταση να στηριχθεί η θέση του Συμβουλίου σε αυτό το θέμα που είναι η μόνη που δεν έχει συμφωνηθεί. Το πρόβλημα είναι πως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη θέση του Συμβουλίου. Κάπως είναι περίπλοκο το πράγμα, αλλά θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Βίκτορ, σε υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να το πετύχω. Το ξέρω. Απλώς θέλω να αναφέρω πως έχει θέση το Συμβούλιο. Κανένα άνοιγμα άλλου θέματος. Και αυτή ήταν και η θέση της, της Επιτροπής και έχοντας υπόψη πως το ΕΛΚΑ επιβεβαίωσε ότι θα επιμείνει στη θέση του Συμβουλίου την προηγούμενη, το οι σοσιαλιστές και οι άλλοι συμφωνούν. Αυτό σημαίνει σαφώς ότι είναι ξεκάθαρη θέση υπέρ της προηγούμενης θέσης του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λάμπερ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω το εξή. Ω εισηγητή και σκέδε εισηγητή, ε, θα πρέπει να πω ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε διαπραγματεύσει ε, ε, προ εξέβρεση συμβιβαστική με το Συμβούλιο. Περίμενα χτε τη συμβιβαστική, το συμβιβασμό, αλλά δεν επετεύθη. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι παρόν, για να τα πω έτσι με δικά μου λόγια, εάν δεν υπάρχει η λύση κοινή, κοινός αποδεκτή δηλαδή, ε, τι μας μένει, μας μένει η θέση του Συμβουλίου και κάποιες φορές αντιμετωπίζουμε προβλήματα, αλλά πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Πρόεδρος. Κλείνω τη συζήτηση, εκτός αν ο εισηγητής θέλει κάτι να πει ακόμα. Ήταν, νομίζω πως τα είπαμε όλοι τι είχαμε να πούμε. Οπότε, εντάξει, προς αυτή την κατεύθυνση μου, όπως συζητάτε. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Επόμενη συνεδρίαση 27-28 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Τέλος της συνεδρίασης.